Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε σιγά σιγά. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Ε, στην ημερήσια διάταξη τώρα προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Σασίλια Μάστρομ, Επίτροπο Αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω ενώπιον μας την κυρία Μάλμστρομ, την Αρμόδια Επίτροπο, με την οποία θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας ε, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Επιτρόπου, έχει τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων, ορισμένα στοιχεία ποινικού δικαίου, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την ε, διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα μας ενημερώσει σήμερα ε, για τα όσα διαμήθησαν στη συνεδρίαση που είχε με τον Υπουργό Αλφάνο ε, της Προεδρίας για το Μάρε Νόστρουμ και το Φρόντεξ. Όσοι ήθιστε, στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο πρώτα οι συντονιστές, η κυρία Μάστον θα απαντήσει και ακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο παρακαλώ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ε, να σας συγχαρώ καταρχήν για την εκλογή σας στη νέα θητεία και εύχομαι να έχουμε αγαστή συνεργασία τους επερχόμενους μήνες μέχρι το τέλος της θητείας. Θα ήθελα να ε, δούμε, να κάνουμε ένα σύνδεσμο μεταξύ της ε, νέας θητείας και της προγενέστερης, προγενέστερης και τα κοινά στοιχεία που μας απασχόλησαν. Γιατί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, το Κοινοβούλιο είναι ισότιμο στις αποφάσεις για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, όπως φάνηκε από τα τελευταία χρόνια συνεργασίας. Θα σας πω πού βρισκόμαστε. Ε, και θα μιλήσω και για ορισμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί για το φθινόπωρο. Ως προς την μετανάστευση και το άσυλο και τα εξωτερικά μας σύνορα, καθώς και την κατάσταση σήμερα, έχουμε να ε, αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση, έκριθμη. Δεν είχαμε ποτέ τόσες σειράξεις παράλληλα μετά τον δεύτερο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και μετά με τόσους ε, πρόσφυγες που υπερβαίνουν τα 52 εκατομμύρια διεθνώς που θέλουν να ξεφύγουν από την καταστολή. Επίσης αντιμετωπίζουμε πολλές σειράξεις, φτώχεια και άλλες δυσχερείς καταστάσεις. Και αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει, καθώς και η Ευρώπη. Ως προς το άσυλο, Ξέρετε ότι η Επιτροπή μαζί με εσάς ενέκρινε το ε, Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου το οποίο είναι αξιόπιστο πραγματικά. Δηλαδή όλοι όσοι αποζητούν άσυλο την χάνουν ίσης μεταχείρισης. Πρόκειται για ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός, αν και θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει και περισσότερο, αλλά δεν στάθηκε δυνατόν. Τώρα θα θέλαμε η εφαρμογή και η μεταφορά να γίνει προς όλα τα κράτη-μέλη, γιατί μόνο έτσι θα είναι λειτουργικό το πλαίσιο και θα ήθελα να πιέσετε τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, είχαμε ανωδική πορεία των ε, προσφύγων και των αποζητούντων άσυλο και αυτό το είδαμε κυρίως στα νότια σύνορά μας. Αλλά οπωσδήποτε και στη Βόρεια Ευρώπη το είδαμε αυτό. Στην Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, εκατοντάδες χιλιάδες ε, μετανάστες προσπάθησαν να ε, περάσουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ευρώπη, δυστυχώς χρησιμοποιώντας σκάφη τα οποία δεν ήταν αξιόπλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση το Mare Nostrum θα πρέπει να επιταχύνουμε το ρυθμό μας όπως απαιτούν ιδιαίτερα οι Ιταλοί. Υποστηρίζουμε τους Ιταλούς ε, μέσα στα πλαίσια του, και του Frontex, πέρα από το Mare Nostrum. Όπως είπε και η Πρόεδρος, ήρθα σε επαφή με τον Υπουργό Αλφάνο την προηγούμενη εβδομάδα και μιλήσαμε για, ένα, για μια επιχείρηση Frontex Plus, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να μας υποστηρίξουν πολλά κράτη-μέλη. Θα μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το πλαίσιο από τον Νοέμβριο δεν είναι αντίγραφο του Mare Nostrum. Ε, πρόκειται για ένα πιο περιορισμένο εγχείρημα, αλλά βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας, γιατί χρειαζόμαστε επιπρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια για αυτή την επιχείρηση, καθώς και πόρους από τον προϋπολογισμό. Ε, ανθρώπινη καταστροφή από τον εμφύλιο στη Συρία, η αστάθεια στο Ιράκ καθώς και στη ευρύτερη γειτονιά μας βλέπουμε ότι ακολουθεί μια πορεία που χρήζει διεθνούς προστασίας. Άλλοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, αλλά πριν από το καλοκαίρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε μία συνεκτική προσέγγιση, δηλαδή επιτάχυνση ε, της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, επέκταση των προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας και προστασίας και καλύτερη ε, δίωξη των ε, εγκληματικών δικτύων καθώς και προστασία όσων χρήζουν προστασία. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις συμβάσεις, καθώς και τις αξίες που δεχόμαστε, αλλά και τη δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης όπως τη γνωρίζουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη μετανάστευση και αυτές οι ροές είναι ευκαιρία και όχι απειλή όπως πολλές φορές απεικονίζεται. Χαίρομαι λοιπόν γιατί έχει επιτελεστεί πρόοδος όσον αφορά την νόμιμη μετάβαση στην Ευρώπη. Και για τους πρόσφυγες μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ε, και για αυτούς που αναζητούν εργασία. Εγκρίναμε την οδηγία για τους εποχικούς εργαζόμενους που είναι το πρώτο νομοθέτημα που αφορά χαμηλές δεξιότητες και τα δικαιώματα των μεταναστών, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Επίσης, μειώσαμε τη γραφειοκρατία μέσα στα πλαίσια των εμπειρογνωμόνων που προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδρασε έτσι ώστε να φτάσει σε ένα εξισορροπημένο κείμενο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την διακυβέρνηση του Σέγγεν. Είχαμε μία προβληματική περίοδο το καλοκαίρι του 2011. Θυμόσαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε επί της ουσίας και ως προς τον τύπο. Αλλά φτάσαμε σε καλά αποτελέσματα. Έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ελεύθερη ε, κυκλοφορία των πολιτών μας και έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης. Όλες αυτές οι αλλαγές ε, έχουν αναγραφεί σε έναν ε, μηχανισμό αποτίμησης του Σέγγεν και αυτό θα κάνουμε και για του χρόνου, την αξιολόγηση που θα γίνει του χρόνου. Επίσης έχουμε ενισχύσει τις πολιτικές σχέσεις με ε, χώρες όπου υπάρχει άρση των θεωρήσεων, ιδιαίτερα με τις πέντε βαλκανικές χώρες και τη Μολδαβία, Περού, Κολομβία και άλλες 17 χώρες. Ελπίζω να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με αυτές τις ε, χώρες πριν από το τέλος του έτους, ενώ η έκθεση αξιολόγησης για την Κολομβία θα εγκριθεί τις επόμενες εβδομάδες για την απελευθέρωση με, ως προς θεωρήσεις με τη Γεωργία, Ουκρανία και Τουρκία επιταχύνονται οι διαδικασίες καθώς και με το Αζερβαϊτζάν ε, και την, ε, την Ισία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και θέματα κινητικότητας. Επίσης, έχουμε συνάψει ορισμένες συμφωνίες επανεισδοχής και αυτό δείχνει ότι λειτουργεί πολύ καλά η πολιτική μας μετανάστευσης και ασύλου. Όσον αφορά την ασφάλεια και τα πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θα ήθελα να μιλήσω για την εμπορία ανθρώπων, κάτι το οποίο ισχύει σε πολλές χώρες. Σήμερα, πέντε χρόνια πριν, υπήρχε διαφορετική προσέγγιση από τα κράτη-μέλη. Άλλοι είχαν ήπια νομοθεσία, άλλοι πιο σκληροί. Τώρα υπάρχει ένα ελάχιστο πλαίσιο διαχείρισης, όπου ε, ακριβώς αντιμετωπίζεται το θέμα χορήγησης ε, βοήθειας ε, ελάχιστης κράτησης και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και ένας συντονιστής ο οποίος συνεργάζεται με τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών και ελπίζω αυτό να σας απασχολήσει και τα επερχόμενα έτη. Ως προς τη διαφθορά είναι μια επιζήμια εγκληματική δραστηριότητα που υποβαθμίζει και την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη δημοκρατία. Στοιχίζει 120 δις ευρώ ετησίως στην Ευρώπη και ίσως η εκτίμηση αυτή δεν είναι σωστή. Η πρώτη έκθεση υποβλήθηκε πέρσι την Άνοιξη και μιλήσαμε για κοινέ λύσεις όπου θα πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες. προσπάθειες. Ελπίζω λοιπόν να δούμε και τις πολιτικές επιπτώσεις αυτής της ε, απόφασης. Επίσης παγώσαμε και κατασχέσαμε έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Το καλοκαίρι ο τύπος ασχολήθηκε με το θέμα της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Υπάρχει η νομοθεσία μας έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε χημικά όπλα υψηλού κινδύνου για να κατασκευαστούν ε, ε, βόμβες και αυτό αφορά και χημικά όπλα, βιολογικά και ούτω καθεξής. Υπάρχει το δίκτυο ε, αντιμετώπισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ένωση των θεμάτων αυτών έτσι ώστε να αποφευχθεί ο βίος εξτρεμισμός. Επίσης, οικοδομούμε πάνω σε αυτή την ε, εμπειρία μας όπου ο ακαδημαϊκός κόσμος, κοιό ε, επικεφαλής ε, θρησκευτικών κινημάτων έχουν δημιουργήσει κομβικά σημεία συνεργασίας. οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ ως προς το PNR, ε, με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, αποτρέπουν την τρομοκρατία. Αυτή την ε, συζήτηση την είχαμε και σε θέματα επαγρύπνησης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να προστατεύουμε και την ιδιωτική ζωή καθώς και τα προσωπικά δεδομένα. Όλα αυτά σχετίζονται και με το, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που αποτελούν πραγματική απειλή και συμφωνήσαμε σε μία νομοθεσία σε σχέση με τις σοβαρές απειλές στο κυβερνοχώρο και η Europol έχει δράσει σε αυτό το τομέα έτσι ώστε να μπορέσει να καταστήλει ορισμένα δίκτυα. Το EC3, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοχώρου, έχει ασχοληθεί και με τους ανηλίκους έτσι ώστε να υπάρξει δίωξη, προστασία των θυμάτων και πρόληψη. Δύο χρόνια πριν, μαζί με τον Αμερικανό ε, Γενικό Εισαγγελέα ασχοληθήκαμε με μια παγκόσμια, ένα παγκόσμιο δίκτυο για την καταπολέμηση του εγκλήματος κατά των ανηλίκων. Και το τελικό σχήμα, θα, μάλλον το σχήμα θα πάρει τελική μορφή τον επόμενο μήνα στην Ουάσιγκτον. Όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε όταν ε, ασχολήθηκε με τις κατευθυντήριες γραμμές τον Ιούνιο, έχουμε επιτελέσει σημαντική εργασία με τους Ευρωπαίους και για τους Ευρωπαίους πολίτες και τώρα θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και θα πρέπει όλη αυτή η νομοθεσία να εγκριθεί, να εφαρμοστεί και να υπάρξει και μία συνέχεια και να δοθεί συνέχεια. Είμαι σίγουρη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο θα συζητήσετε και θα ασχοληθείτε με την χρηματοδότηση, ίσως και σε ένα απότερο στάδιο. Και ε, ο συνεργάτης θα σας παρουσιάσει τις λεπτομέρειες. Η επόμενη επιτροπή θα ασχοληθεί με νέες πρωτοβουλίες, αλλά πριν ε, απαλλαχθείτε από μένα, Έχουμε ορισμένα ζητήματα επιτάπητος, ε, τα οποία θα μας απασχολήσουν άμεσα. Η ε, μεταρρύθμιση της Europol, βλέπω τον Αγκουστίν μπροστά μου, καθώς και την ε, προσέγγιση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το φθινόπωρο. Η Europol θα γίνει πιο λειτουργική ε, τηρώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων. Επίσης, θέλουμε να ε, λισαβονοποιήσουμε τη ΣΥΠΟΛ και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εγκαίρως, διότι έτσι θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το ε, σχήμα, με το σχέδιο μάλλον κατάρτισης για την ε, πραγματική χρήση όλων αυτών των σχημάτων. Επίσης, το προσωπικό της ΣΥΠΟΛ θα είναι σίγουρο για το μέλλον του οργανισμού. Επίσης, θα θέλαμε ε, ε, να ασχοληθούμε και με την κατάρτιση. Η Σεσίλια Βίκστρομ έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά ως προς το, τους φοιτητές και τον ακαδημαϊκό κόσμο, κατάρτιση και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι νέοι να συνεισφέρουν με τις, ε, ε, με τις μελέτες τους και ως προς το πακέτο των θεωρήσεων θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τρίτες χώρες καθώς ε, και στα πλαίσια των ε, προξενείων που θα εκδίδουν θεωρήσεις βάσει συμφωνίας Σέγγεν. Επίσης, το καλοκαίρι είχαμε την ε, επίσημη συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το PNR. Υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας ε, το οποίο έχει επιτελέσει πρόοδο σε σχέση με τις ρήτρε διασφάλισης προσωπικών δεδομένων. Ελπίζω να το εγκρίνετε στο μέλλον. Μιλώντας για PNR, Τις τελευταίες ημέρες ε, είδαμε τρομακτικές εικόνες από το Ιράκ και τη Συρία και αυτό έχει επίπτωση και στα δικά μας κράτη στα πλαίσια του ε, Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων ασχοληθήκαμε με τους ξένους μαχητές που αποτελούν πραγματική απειλή για την Ευρώπη. Πρόκειται για Ευρωπαίους υπηκόους που συμμετέχουν σε αυτές τις διεθνείς σειράξεις και λαμβάνουν και όπλα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα, γι' αυτό θα ήθελα ο κύριος Κύρκο, ο εισηγητής, να ασχοληθεί την με τις να συνεχίσει τις εργασίες του ως προς ένα ευρωπαϊκό PNR. Αυτά ήθελα να πω σε όλους και ιδιαίτερα στα νέα μέλη για να ξέρουν πού βρισκόμαστε. Όλοι έχετε δεσμευτεί σε αυτά τα ζητήματα, αν και πολλές φορές διαφωνούμε για την αντιμετώπιση τους, ως προς την αντιμετώπιση τους, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω σχόλια και να απαντήσω και τις υπόλοιπες εβδομάδες συνεργασίας ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία ε, Μάστρομ, κυρία Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί διατελέσατε και ευρωβουλευτής και ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, οι συντονιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, κυρία Μέτσολα. Έχουν γίνει μεγάλες βελτιώσεις στο θέμα που σας απασχολεί ιδιαίτερα σπαστικοποίηση και ε, ε, την ε, τρομοκρατία. Εγώ θα μιλήσω για την παράνομη μετανάστευση, το Frontex SIN ή την επιχείρηση Τρίενα. Εγώ είμαι από τη Μάλτα. Ξέρω πόσο σημαντικό ήταν το Μάρε Νόστρομο σε επιχείρηση διάσωση ζώων και στο μέλλον θα πρέπει να έχει την επαρκή υποστήριξη για να έχει άλλα αποτελέσματα. Επίσης, ε, όταν αρχίσατε αυτή την επιχείρηση είπατε ότι θα πρέπει να περάσουν τα κράτη-μέλη από την προφορική αλληλεγγύη στην έμπρακτη πλέον ε, και με το χέρι στην τσέπη. Συμφωνώ απολύτως. Ε, κάποια όμως ε, δημοσιεύματα μου φαίνονται αρκετά ασαφή και συγκεχημένα. Ορισμένοι λέγουν ότι θα αντικαταστήσετε το Μάρε Nostrum, ότι θα το συμπληρώσετε, ότι θα το υποστηρίξετε. Τι θα κάνετε. Χρειάζεται καλύτερα να μας ε, διευκρινίσετε και να ορίσετε τι θα γίνει. Πάντως είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε επιχείρηση χρειάζεται την υποστήριξη των κρατών μελών και ε, σε δυναμικό και οικονομικά και ε, σε στελέχη, αλλιώς θα αποτύχει αυτή και η Frontex ίδια. Μπορείτε να μας πείτε πώς αντέδρασαν τα κράτη-μέλη, να μας το πείτε σήμερα αυτό. Και τέλος να σας ευχαριστήσω και πάλι και ε, θέλω να σας δω και αύριο στην έδρα της ΕΙΑΣΟ, του Γραφείου για το Άσυλο. Ευχαριστώ η κυρία Ζήπελ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η προλαλή σας θα σας ήμουν ευγνώμων κυρία Μάλστρομ αν μας εξηγούσατε λίγο περισσότερο ε, πώς θα λάβει σάρκα και οστά αυτή η επιχείρηση Frontex Plus, Frontex Sin. Ακούμε ότι θα αρχίσει το Νοέμβρη. Τα κράτη-μέλη όμως τι κάνουν και με ποιο τρόπο συμμετέχουν. Και θα με ενδιαφέρει και μια άλλη ερώτηση, διότι εδώ δεν μας ενδιαφέρει μόνο η διάσωση των ε, προσφύγων, αλλά εγώ διαρωτώ με Μήπως έχει την πρόθεση η Ιταλική κυβέρνηση οι πρόσφυγες αυτοί που διασώζονται στα χωρικά ύδατά τους να μην παραμένουν όλοι στην Ιταλία. Υπάρχουν σχέδια βέβαια να σώζονται οι άνθρωποι αυτοί, αλλά σε αντίθεση με τα όσα συνέβαιναν μέχρι τώρα να ε, ε, ε πηγαίνουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Και θέλετε να συνενώσετε και κάποιες άλλες δράσεις, ερμής και μια άλλη για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά στα ίδια τα σύνορα και μεσοπέλαγα ποιος αποφασίζει ε, κάποιον άνθρωπο αν είναι παράνομος μετανάστης ή αν είναι πρόσφυγας που δικαιούται άσυλο. Επίσης αναφερθήκατε στην νόμιμη μετανάστευση γιατί όντως πολλοί προσφυγέ είναι οικονομικοί μετανάστες που θέλουν να δουλέψουν σε εμά. Τι γίνεται με την μπλε κάρτα και με την ε, οδηγία για τους εποχικούς εργαζομένους. Υπάρχει δυνατότητα εκεί να αυξηθεί, σχεδιάζεται τίποτα για την αύξηση της νόμιμης μετανάστευσης. Και επίσης, οι άνθρωποι αυτοί από τις τρεις χώρες γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν τέτοιοι νόμιμοι τρόποι και τους χρησιμοποιούν. Και ένα τελευταίο για τους λεγόμενους ξένους μαχητές foreign fighters. Εδώ γιατί χρειάζεται PNR και με ποια αιτιολόγηση απαγορεύει κάποιος ένα Γερμανό ή θέλει να απαγορεύσει κάποιος ένα Γερμανό που επιστρέφει από τη Συρία να εισέλθει στη Γερμανία. Εσείς έχετε στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λέει, μια χώρα ένας αριθμός μέχρι 300. Πώς, βρίσκεται αυτός ο αριθμός. Τους γνωρίζουμε και αν τους γνωρίζουμε γιατί δεν τους ασκούμε ποινική δίωξη. Απλώς υποθέτουμε ότι έχουν πάει στη Σύρια για να ε, πολεμήσουν και είναι γύρω στους 300 από την τάδε χώρα. Υπάρχουν ε, και δικαιώματα δικονομικά και υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Και εγώ θέλω και τέτοιες οδηγίες να δω. Δεν μπορούμε να εκδίδουμε ανθρώπους, να τους απελάβνουμε, να τους παίρνουμε τα διαβατήρια, να τους αφαιρούμε την ηθαγένεια, απλώς και μόνο επειδή υποπτευόμαστε, υποθέτουμε ότι έχουν διαγωγή κοσμία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύρκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, η συνείδηση αγωγής θέλω να καταγραφεί πως είμαστε γνώμονες προς την Επίτροπο. Ε, πήρε μόνο λίγα στοιχεία από το σημείωμά της, αλλά ε, δείχνει πόσο σημαντικές, ε, πόσο τεράστιες είναι αυτές οι προκλήσεις ε, που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και θα ήθελα όχι μόνο να εκφράσω τις ευχαριστίες μας, αλλά να την ευχαριστήσω για την προσέγγιση ε, που υιοθέτησε για όλα αυτά τα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει. Ήταν εξαιρετική ε, η προσέγγιση και ο τρόπος που τα χειρίστηκε. Ε, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με το έργο σας. Αυτά. τώρα, έχω τρία-τέσσερα σημεία να θέσω. Θα είμαι σύντομος. Δεν θέλω τώρα να αρχίσουμε με το PNR γιατί θα βαρεθείτε όλοι. Ξέρετε, τώρα κλαίνει ο καθένας το δικό του και τίποτα δεν γίνεται. Νομίζω ότι ε, για τους freedom fighters, ε, για τους ε, μαχητές, από αυτά που είπατε και για την κατάσταση ασφάλειας προκύπτει με σαφήνεια, αν δούμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ότι πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα αυτό το θέμα. Εγώ θα βάλω τα δυνατά μου και ελπίζω να πείσω και τους συναδέλφους για να το προωθήσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια πάντως για την εμπορία ανθρώπων, ε, ε, εμένα με ανησυχούν τα παιδιά. Τα παιδιά, η εμπορία των παιδιών ε, είναι ντροπή και έσχος αυτό που συμβαίνει από ηθικής πλευράς, πέρα από το ότι είναι μια εγκληματική πράξη. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να γνωρίζουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις και λυπάμαι που το λέω, την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισης όπως και οι ενήλικες ως προς την υποδοχή, την ε, φύλαξη, την ε, ε, σύλληψη ορισμένες φορές. Μα πού είναι η ανθρωπιά μας, πρόκειται για παιδιά, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, μόνο και μόνο για τη φήμη, για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά. Πριν αρχίσει η συνεδρίαση αυτό συζητούσαμε κάποιον για, σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας. Θα συμφωνήσετε νομίζω ότι στο νέο γύρο, γιατί με μέρη εισηγητής για το, τα όσα κάνουμε για το ξέπλυμα αυτή τη στιγμή, ε, ελπίζω να εστιάσετε την προσοχή σας στην αναλογικότητα, να ασχοληθείτε με τους πραγματικούς μεγάλους εγκληματίες, ε, δράστες, αυτούς που ε, νομιμοποιούν παράνομα έσοδα σε μεγάλη κλίμακα ε, και ταυτόχρονα αυτοί που λειτουργούν σύνομα και ε, μεταχειρίζονται αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να σφερόμαστε ανθρωπινά. Ε, τώρα σε σχέση ε, με την Μεσόγειο, την Task Force, το Ταμείο Ένταξης, ΕΑΣΟ, Frontex, ναι έχουμε διαθέσει αυξημένα κονδύλια όμως είναι σημαντικό με αυτά τα χρήματα ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να ε, ξεκαθαρίσουν, να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι ο ρόλο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ορισμένε φορέ οι πρόσφυγε και οι ετούντε άσυλο την χάνουν χείρι τη μεταχείριση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είπατε κι εσεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ει δρόμου μεταναστών προ την Ευρώπη. Οι κανόνε είναι κανόνε όμω και οι καταχρήσει είτε από εγκληματικέ οργανώσει είτε από άτομα είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχόμαστε και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από την πραγματική προτεραιότητα, ε, δηλαδή να προστατεύσουμε τους πραγματικούς, ε, τους γνήσιους ε, πρόσφυγες και του άσυλο και αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν στο ιστορικό της Ευρώπης, όχι για να καταχραστούν τους κανόνες, αλλά για να εργαστούν. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Κίρχοπ Βίκστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την ε, τραγωδία ξέρουμε όλοι τι συνέβη πριν από ένα χρόνο περίπου και όλοι οι ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέφρασαν τη λύπη τους, ε, απέφτυναν έκκληση για ανάληψη άμεσης δράσης, πραγματικά ορισμένοι φορτώνουν το βάρος και την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα ίδια κράτη-μέλη πάντοτε παρεμποδίζουν τις πρωτοβουλίες σε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ξέρουμε. Ο Frontex δεν έχει πόρους ε, και δικό του εξοπλισμό οργανισμός και η επιτυχία λοιπόν της επιχείρησης Frontex είναι ε, ε, εξαρτάται απόλυτα από τη βούληση των κρατών μελών να συμβάλλουν στις επιχειρήσεις μεταξύ άλλων διάσωσης ανθρωπίνων ζώων. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των κρατών μελών. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα το ανακοινωθέν της 27 Αυγούστου. Λοιπόν, μόλις ανακοινώσατε στην επιχείρηση Frontex είναι. Ποιε αντιδράσει υπήρξαν από πλευρά των κρατών μελών και είναι συμπληρωματική η επιχείρηση σε σχέση με τη Mare Nostrum και θα συνεχίσει η Mare Nostrum να, να ε, διεξάγεται αυτή η επιχείρηση. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Ο Frontex επίση ε, θα αρχίσει να αναλαμβάνει επιχειρήσει διάσωση. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ε, Τέλο, πότε θα είναι διαθέσιμο για μα εδώ στην Επιτροπή το επιχειρησιακό σχέδιο του Frontex Sin για να δούμε τις δικλείδες ασφαλείας, παραδείγματος χάρη, ως πρόσφερη πίνη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο μέτρο του δυνατού θα πρέπει να συμμετάσχουμε στη διαδικασία, διότι μην ξεχνάμε ότι και εμείς συμμετείχαμε στην τροποποίηση του κανονισμού Frontex και προσθέσαμε σημαντικότατες ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άρα ε, θα ε, χρειαστεί με μεγάλη προσοχή να μελετήσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο του Frontex. Έχω και πολλά άλλα να πω, αλλά θα ε, συγκρατηθώ διότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν και θα συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε. Ernst. Ευχαριστώ. Τρία θέματα. Πρώτον, για να εμβαθύνουμε λίγο. Ε, άσυλο και μετανάστευση φυσικά. Έχουμε τεράστια ρεύματα αυξανόμενα μεταναστών, τα είπατε και είναι γεγονός αυτό ισχύει. Και το ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη περισσότερο και ιδιαίτερα για τους ετούντες άσυλο. Είπατε για το Mare Nostrum ε, που αντικαθίσταται τώρα από το Frontex ε, Plus ή SIN και μια επιπλέον προσπάθεια. Ωραία, ερωτώ εγώ. Και ποιο είναι το κόστος. Είναι τελείως ασαφές. Το έχετε υπολογίσει. Έχετε καμιά ιδέα, τάξη μεγέθους, για ποια ποσά μιλάμε. Και μετά έχουν δεσμευτεί διάφορα κράτη-μέλη να βοηθήσουν. Ποια έχουν δηλώσει ήδη προθυμία. Και ένα τρίτο. Η επανεγκατάσταση. Resettlement. Πώς το έχετε σκεφτεί, έχετε προβλέψει κάποια μέτρα, κάποια κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα ειδικό αυτό και ποιο ρόλο θα ε, παίξουν εκεί οι κατευθυντήριες γραμμές για ε, τη διάσωση στη θάλασσα. Και πώς θα αξιολογείται η αίτηση ασύλου και θα προωθούνται σε τρίτες χώρες οι άνθρωποι αυτοί. Ένα δεύτερο, οι τζιχαντιστές που ε, αναφέρθηκε επανειλημμένα αυτό το θέμα. Ότι πρόκειται να αλλάξουν εξαιτία του οι κανόνες εισόδου και εξόδου από τις χώρες. Ε, εγώ καταλαβαίνω τη βασική ιδέα που κρύβεται από πίσω, αλλά στο δίκαιο η κατάσταση έχει ω. εξή. Όταν ανοίγω μια πόρτα μπορούν να περάσουν διάφορα. Και μπορεί να αρχίζει από του τζιχαδιστέ και αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλου προσοχή να δούμε τι θα κάνουμε ουσιαστικά και πραγματικά με αυτή την ομάδα ανθρώπων. Τα είπε και η κυρία Ζίπελ. Νομίζω ότι εδώ ανοίγουμε πόρτες ε, και θα το μετανιώσουμε στο μέλλον. Και το τρίτο και κύριο και δεν θα σας εκπλήξει, μιλήσατε για το PNR, τα δεδομένα των επιβατών και ενθουσιάστηκε και ε, ο κύριος Κίρκοπ. Δεν χωράει καμία αμφιβολία, καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά για την προληπτική διατήρηση και ε, αποθήκευση δεδομένων. Αυτό θεωρήθηκε άκυρο και ως μη γενόμενο. Και η ίδια η οδηγία ολόκληρη επεφάνθη το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και άμα διαβάσετε προσεκτικά την απόφαση, τι λέγει. Ξεκάθαρα και μόνο από το γεγονός ότι αφορά αυτό όλο τον πληθυσμό γενικά και αδιάκριτα και όλα τα στοιχεία, κάνουμε και μια τρύπα στο νερό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οπότε αυτή η προληπτική διατήρηση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων ε, και αυτή η απόφαση τι επιπτώσεις έχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλάζουν κανονισμοί, οδηγίες, έχετε εσείς ενέργειες ε, προς την κατεύθυνση αυτή ε, ε, αναλάβει. Και σε εθνικό επίπεδο φαντάζομαι θα πρέπει να συμβούν όλα αυτά. Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για να τα εξετάσετε ή τι προτίθεστε να κάνετε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτά. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Δύο συντονιστές ακόμα έχουμε. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να στραφώ στο Μάρε Νόστρομ, αλλά θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Μιλήσατε για πολλές χώρες, αλλά δεν μιλήσατε για το κοσυφοπέδιο. Ως προς το Μάρε Νόστρομ, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το Frontex Plus ε, θα αντικαταστήσει το Mare Nostrum. Επίκειται κάτι τέτοιο. Εάν όχι, ποια τμήματα δεν θα παραμείνουν καλυμμένα ως προς τη Μεσόγειο. Δηλαδή, πού θα πούμε, α, εδώ θα αφήσουμε τους ανθρώπους να πεθάνουν. Το θέμα δεν είναι ίσονο σημασία. Σε πάση περιπτώσει θα ήθελα να αναρωτηθώ κατά πόσο η Frontex μπορεί να αντιμετωπίσει και να αντικαταστήσει το Mare Πρόκειται για έναν οργανισμό που ασχολείται με την φύλαξη των συνόρων. Εμείς χρειαζόμαστε μία ανθρωπιστική ε, αποστολή στη Μεσόγειο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιζήσουν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της Frontex. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και δεν καταλαβαίνω πώς ένας οργανισμός διαφύλαξης των συνόρων μπορεί να μετατραπεί σε έναν ανθρωπιστικό οργανισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και θα ήθελα να ε, θέσω τις αμφιβολίες μου επί του θέματος. Και έχω και άλλες ερωτήσεις ως προς τις λεπτομέρειες. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτούς τους οποίους ε, μπορούμε να περισσώσουμε. Ποιος θα αναλάβει, πώς θα έχει ο επιμερισμός ευθυνών σε σχέση με τη Frontex και πώς ε, θα είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε τους πάντες, όχι μόνο τους παράνομους. Ποιος θα αναλάβει την διαχείριση των κέντρων διαβίωσης. Είδαμε πολλές φορές ότι ε, αντιμετωπίσαμε τραγωδίες γιατί δεν ήταν σωστές, σωστά επιμερισμένες, επιμερισμένες οι ευθύνες. Και ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της συγχώνευσης, τη στιγμή που οι στόχοι είναι διαφορετικοί και ποιες θα είναι οι δραστηριότητες της ε, Frontex ε, Plus, δηλαδή ένα αέρια παρακολούθηση, θαλάσσια, τι. Ως προς τον προϋπολογισμό είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο τμήμα του προϋπολογισμού της Frontex θα αποδοθεί στη Frontex Plus τι απαιτείται από τα κράτη-μέλη ως προς προσωπικό ή εξοπλισμό καθώς και χρηματοδότηση, διότι η Ιταλία ανέφερε ότι αν είναι ε, χώρα υποδοχής θέλει και χρηματική αποζημίωση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει η Frontex διαβάσαμε στο γερμανικό τύπο ενδιαφέροντα ε, στοιχεία από τη γερμανική και ιταλική κυβέρνηση που συνεργάζονται με τη γαλλική για μια νέα ε, πρωτοβουλία επιμερισμού ευθυνών. Είπαν ότι θα πρέπει το μοίρασμα να είναι διαφορετικό κάτι το οποίο είναι και κάπως αντιφατικό. Δεν ξέρω αν ακούσατε για αυτή την πρωτοβουλία και τι σημαίνει αυτό για το Δουβλίνο 3. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φεράρα είναι η τελευταία συντονίστρια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρία Μάλστρεμ. Μάλλον θα επαναλάβω ε, πολλά πράγματα γιατί θα πω αυτά που προείπαν αρκετοί συνάδελφοι. Σε τι διαφέρει το Frontex Plus σε σχέση με το Μάρε Νόστρουμ, διότι ο Υπουργός Εσωτερικών ε, Αλφάνο ε, λέει ακριβώς ότι η Frontex Plus θα αντικαταστήσει το Mare Nostrum, αλλά το περιεχόμενο είναι διαφορετικό. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Πού διαφέρουν αυτά τα δύο σχήματα. Η Frontex ε, Plus δεν θα ασχοληθεί και με τα διεθνή χωρικά ύδατα. Θα διαφέρει από το Mare Δηλαδή τι θα γίνει με τα ε, σκάφη τα οποία βρίσκονται σε διεθνή χωρικά ύδατα. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται σε διεθνή χωρικά ύδατα. Δηλαδή τι κάνουμε, ε, εποπτεύουμε τα σύνορα, πώς ορίζουμε την βοήθεια, την έμπρακτη βοήθεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας που οριζόταν από το Mare Nostrum που λύγει το Νοέμβριο. Ίσως και η Γαλλία και η Γερμανία προσχωρήσουν. Τα άλλα κράτη-μέλη τι θα κάνουν. Δεν θα φέρουν καμία ευθύνη. Ποιος θα είναι ο ρόλος τους στα πλαίσια αυτής της επίγουσας βοήθειας για τη μετανάστευση. Μιλάμε για 83 εκατομμύρια, 32 εκατομμύρια για την ενοικίαση και ούτω καθεξής. Μιλάμε για τα έξοδα της Frontex. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερα να προβλέψουμε μία έδρα, την έδρα στη Σικελία, γιατί η Σικελία κατακλείζεται από αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Η Άζο θα μπορούσε να ασχοληθεί περισσότερο στην Ιταλία, διότι εμείς λαμβάνουμε το 60% των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου. Ευχαριστούμε κυρία Φεράρα. Επίτροπε, ακούσατε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα σας δώσω το λόγο για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω όλοι αναφερθήκατε στο Frontex και στη Mare Nostrum. Θα αρχίσω από αυτό λοιπόν και εγώ. Ε, πάντως, αν δεν κάνω λάθος, ε, αύριο το πρωί θα έχετε τον αναπληρωτή ε, Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Χιλάρια, και μπορεί να σας απαντήσει για τα τεχνικότερα ζητήματα. Ε, μετά την ε, τραγική καταστροφή στην Λαμπεντόσα ε, άρχισε αυτή η Ιταλική, αμυγός Ιταλική επιχείρηση Mare Nostrum. 100.000 άνθρωποι έχουν σωθεί νομίζω από το Ιταλικό ναυτικό. Είναι εξαιρετική και άνευ προηγουμένου αυτή η επιχείρηση και συγχαίρω τους Ιταλούς. Είναι πραγματικά καταπληκτικό αυτό που κατάφεραν. Βέβαια η τραγική άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι αυξήθηκε η ένταση των εισδροών από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Δηλαδή ε, είναι ακόμη μικρότερες ε, οι λέμβοι, ακόμη περισσότεροι άνθρωποι πάνω σε αυτές τις λέμβους, ακόμη λιγότερο ε, ασφαλή τα σκαφίδια στα οποία μεταφέρονται οι άνθρωποι και πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό ε, το θέμα. Τι συμβαίνει τώρα με τη Μαρινόστρουμ, είναι ιταλικό το ζήτημα, δεν έχουμε άποψη εμείς γι' αυτό, γίνονται συζητήσεις στην Ιταλία, αλλά είναι θέμα της Ιταλίας στο μέλλον του Μαρινόστρουμ. Ξέρω ότι υπάρχει μια πρόθεση τροποποίησης της επιχείρησης και σταδιακής εξάλληψη. Ναι, ε, αλλά μέχρι εκεί. Ε, Frontex είναι, έτσι ε, έχουμε ονομάσει το πρόγραμμα προ το παρόν. Δεν ε, ισούται με το Mare Nostrum. Δεν έχουμε ε, τις δυνατότητες, το προσωπικό, την εντολή, τα λεφτά, τους πόρους για να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κοστίζει πάρα πολύ το Μαρινόστρουμ. Ο Frontex αποκλείεται να αναλάβει κάτι τέτοιο και το έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πολύ καιρό τα κράτη-μέλη. Δεν γίνεται να αντικαταστήσουμε εμεί το Μαρινόστρουμ. Μπορούμε να το συμπληρώσουμε και ε, να είναι πιο περιορισμένη κλίμακα η επιχείρηση. Συνεργαζόμαστε με τι Ιταλικέ αρχέ και ε, ελπίζουμε και με τι ε, Μαλτέζικε για... και στη συνέχεια και άλλε χώρε ελπίζουμε για να προσδιορίσουμε από κοινού το εύρο και την εμβέλεια τη επιχείρηση χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία, αποτίμηση του κόστους, ε, του προσωπικού που χρειάζεται, σκάφη, ελικόπτερα, ε, γενικότερα υλικοτεχνική δυνατότητα. Πρώτα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και μετά μπορώ να είμαι σαφέστερη, αλλά ε, τις ερχόμενες ημέρες, εβδομάδες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας, σίγουρο είναι θα είναι πιο περιορισμένη η επιχείρηση, διότι η εντολή του Frontex, όπως ξέρετε, είναι όποιος κινδυνεύει συνέβη τον σώζουμε. Ε, όπως είπε η κυρία Σίπελ και άλλοι, ε, είναι ε, συνοριοφύλακες ουσιαστικά, τίποτα παραπάνω. Ε, ε τώρα, ε, όλο ένα και περισσότεροι θα προσπαθούν ε, να περάσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη. Είναι φοβερές οι σειράξεις γύρω-γύρω, ακόμη και λίγοι να έρθουν από τη Συρία. Ε, προς την Ευρώπη ε, δεν, ε, θα δεν μπορεί να σταματήσει αυτή η ροή αν θέλετε η μεταναστευτική και δεν έχουμε λύση έτοιμη να σας την πούμε. Σφαιρικά πρέπει να το δούμε το ζήτημα. Φυσικά τους καταβλισμούς προσφύγων εκτός Συρίας πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Η Επίτροπο Διοντζίβα ασχολείται με το Ιράκ και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε και εκεί το ίδιο και σε σχέση με την εμπορία ε, ανθρώπων με τις ε, χώρες ε, διέλευσης, όπου είναι αυτό δυνατό, έτσι, την Ισία. με τη Λιβύη πάλι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Ε, να φροντίσουμε να λαμβάνεται υπόψη η κείμενη νομοθεσία, οι συνθήκες υποδοχής να είναι ίσες, ε, όλα τα κράτη-μέλη να επομίζονται τις ευθύνες τους, ώστε να είναι δίκαιη η εξέταση ε, του φακέλου τους, να σέβονται τη διαδικασία του Δουβλίνου. Κυρία Σίπελ, καλά τα είπατε. Όποιος ζητάει το άσυλο δικαιούται εξέταση του φακέλου του ενδεχομένως θα χορηγηθεί ή και όχι. Ε, αλλά στη συνέχεια αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να εφαρμοστεί ε, σωστά η οδηγία ε, για το άσυλο και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι υπερβολικά χρονοβόρα η διαδικασία. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε. Η απόδοση των ανθρώπων είναι έγκλημα και αυτό παραβιάζει και τη δική μας νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Η εξώθηση των ανθρώπων είναι παράνομη, συμβαίνει συμβαίνει. Ναι, συμβαίνει παντού στην Ευρώπη, αλλά κάθε φορά που γίνονται καταγγελίες εμείς προσπαθούμε να αναλάβουμε μέτρα και να ζητήσουμε έρευνα ε, να γίνει από τα ε, ε, καστοτε κρατη κράτη-μέλη και ανάληψη των προσφορότερων μέτρων. Τώρα πόσο θα κοστίσει αυτό, τι να σας πω. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε πιστώσεις από τον φετινό στον προϋπολογισμό του 2015 να συγχωνεύσουμε κόστος, πώς το λένε, α ναι, το τον Ερμή και τον Ενέα ε, για να, ε, να καθαρίσουμε τον προϋπολογισμό, να συγχωνεύσουμε τις δύο επιχειρήσεις και να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση κονδυλίων, να έχουμε κοινά, κοινούς πόρους ε, αλλά και περισσότερα κονδύλια. Ε, και πρέπει να παίξετε και εσείς το δικό σας το ρόλο, γιατί και εσείς να αποφασίσετε για τον προπολογισμό. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο πρέπει να πιέσετε όταν είναι ξεκάθαρε, οι αρμοδιότητε, ε, η εντολή και τα, τα καθήκοντα του Frontex και θα γίνει αυτό, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλώ δεν έχει γίνει, ε, να επιμείνετε και αύριο το πρωί ο σε Γενική Διευθυντή ε, θα σα μιλήσει περισσότερο για τα τεχνικά ζητήματα. Τότε θα συζητηθούν ε, τα πράγματα μεταξύ κρατών μελών και εμείς ε, με τον Ιταλό Υπουργό Αλφάνο θα αρχίσουμε τις διμερείς με τα κράτη-μέλη για να δούμε. Έχω ήδη κάποιε ενδείξει. Η Γαλλία παραδείγματο χάρη προσφέρει την υποστήριξή τη. Ο κύριο Αλφάνο ταξιδεύει αυτή τη στιγμή και εγώ στη Μάλτα θα πάω αύριο γιατί είναι από του άμεσα η λειτουργία τι γίνεται με τους ε, ε, ανθρώπους που σώζουμε. Αυτό ε, θα ξεκαθαριστεί πρωτού αρχίσει η διαδικασία. Με τους υπουργού. θα συζητήσουμε για τον επιμερισμό των βαρών. Δεν μου αρέσει να λέω των βαρών γιατί είναι επιμερισμό των ευθυνών και όχι των βαρών. Δεν είναι βάρος οι άνθρωποι. Σήμερα 5-6 κράτη-μέλη υποδέχονται σχεδόν όλους τους πρόσφυγες. Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Δανία ε, μετά από την Ιταλία υποδέχονται το 75% των ετούντων άσυλου Μετά έρχεται το Βέλγιο ε, και ε, έχουμε περίπου 15 κράτη-μέλη που δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Είμαστε 28 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τόσες ε, χώρες με τις οποίες γειτονεύουμε, δεν κάνουν τίποτα. Μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, όχι. Μπορούμε να τους πιέσουμε, να εφαρμόσουμε τους κανόνες, όχι η απάντηση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε, να ε, συμμετέχουν σε προγράμματα επανεγκατάστασης, τους πλέον ευάλωτους δηλαδή θα τους ε, πάρουμε από αυτή την περιοχή ε, και έχουν υπάρξει κάποιες ευελτιώσεις αλλά ε, σε πολύ μικρό βαθμό διότι ε, γιατί, γιατί έρχονται παράνομα στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι, γιατί νόμιμος τρόπος δεν υπάρχει. Πρέπει να το βρούμε και αυτό. Πολύ λίγα γίνονται σε αυτό το τομέα. Ε, η κλίδα κατανομής, ε, ε, όλα τα think tanks συγκεντρώνουμε όλες τις ακαδημαϊκές μελέτες για να έχουμε τα στοιχεία είναι εφικτό αυτό, αλλά προς το παρόν από κάποια κρατημέλη έχουν πολύ, γίνει πολύ λίγα. Μπορεί να αλλάξει αυτό και ο διάδοχός μου μπορεί να καταφέρει περισσότερα πράγματα. Στις 8-9 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο θα ξανασυζητηθεί το ζήτημα. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα αυτό το ζήτημα, αλλά όλοι με ρωτάγανε γι' αυτό. Ε, μπορώ, μπορώ να απαντήσω, αλλά προτιμώ να έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου. Για τους ξένους μαχητές συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ε, 9 με 10 χώρες στην Ευρώπη έχουν δηλώσει ότι οι δικοί τους ε, υπήκοοι οι πολίτες έχουν πάει στο Ιράκ ε, με το Ισλαμικό κράτος ή άλλοι. Ε, άλλοι φεύγουν. Ε, εκείνος ε, που σκότωσε τέσσερις στο Εβραϊκό Μουσείο το Μάιο ε, ε ήταν τέτοιος ξένος μαχητής. Και ε, έχουμε και στην Νορβηγία και στη Σουηδία και στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Πρόκειται για συνεργασία αστυνομία και μυστικών υπηρεσιών. Δεν έχουμε ε, τη δυνατότητα να επιβάλλουμε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία ποιος δύναται να εισέρχεται, να εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να ε, του κατάσχεται το διαβατήριο. Δεν είναι κοινοτική νομοθεσία, είναι αμυγός ε, εσωτερικά θέματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθίσουμε μαζί, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να έχουμε το δίκτυο αυτό το ραν ε, ε, συνειδητοποίησης της για να συνεργαστούμε να δούμε με ιδέες πώς μπορούμε να ε, κοιτάξουμε τα θύματα, ε, πώς ε, με κάποιους που επιστρέφουν μετανοημένοι τέτοιοι μαχητές να συνεργαστούμε. Υπάρχουν δυνατότητες για ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι εκεί όμως η συνεργασία. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Κίρκοπ. Για το, η διακίνηση ανηλίκων είναι πραγματικά ένα δραματικό θέμα και με τη μετανάστευση, όταν αυτό συνδέεται, έχουμε ειδικέ διατάξεις και πρόνοιες για να προστατεύονται οι ανήλικοι, ενώ ιδιαίτερα όταν πρόκειται ε, για καταναγκαστική παιδική εργασία ή για σεξουαλική κακοποίηση, ε, προβλέπονται αυτά στην αντίστοιχη οδηγία, αλλά βεβαίως θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Νομίζω το παρακολουθεί ο κύριος Μπαρνιέ και κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το τομέα ο συνάδελφος και σας παραπέμπω σε εκείνον. Για το Κόσοβο, ναι δεν το ανέφερα, είναι η μόνη χώρα στα Βαλκάνια με την οποία Δεν έχουμε ακόμα απελευθερώσει τις θεωρήσεις, έχουμε συνεργαστεί βέβαια μαζί τους. Μας κατέθεσαν για δεύτερη ε, εκτίμηση και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του θέρους. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Τώρα ξέρετε ότι είναι και σε διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν γίνονται πολλές συζητήσεις, αλλά οι βελτιώσεις είναι πολύ σημαντικές και Έχουμε και άλλες συστάσεις ε, για ε, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ένταξη ε, επαναπαρατηθέντων και θέματα εγκλήματος και διαφθοράς. Συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας και αυτή τη στιγμή συμμετείχε η κυβέρνηση θα συνεχίσουμε. Ο στόχος είναι βεβαίως κάποια στιγμή να μπει και το Κόσοβο στις χώρες ε, που δεν χρειάζονται θεώρηση διαβατηρίων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως μέχρι ε, να καλυφθούν, να πληρωθούν όλα τα κριτήρια. Τελευταίο για την διατήρηση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Φαντάστηκα ότι θα με ρωτούσατε. Ήρθε το δικαστήριο και απεφάνθη ότι η οδηγία αυτή, όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αναλογική. Αυτό συμφωνεί πάρα πολύ με την αξιολόγηση που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μια διετία, που είχε επικρίνει την ισχύουσα οδηγία για πολλά ζητήματα το δικαστήριο δεν λέγει ότι η συλλογή στοιχείων και δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος ε, απαγορεύεται. Να είναι αναλογική λέει και αποφαίνεται ότι η οδηγία δεν είναι αναλογική, αλλά όχι ότι απαγορεύεται. Η εθνική όμως νομοθεσία δεν εμπίπτει ή δεν καλύπτεται από την απόφαση αυτή απαραίτητο. Θα πρέπει τα εθνικά δικαστήρια να το εξετάσουν. Βεβαίω το να λύουμε με τους νομικούς μας έμπειρογνώμονε είναι περίπλοκο αρκετά. Τώρα θα υπάρξει νέα πρόταση πιο περιορισμένη, είναι πολύ νωρί να το πούμε. Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιληφθεί και θα το συζητήσει σε συνεργασία μαζί σα για να αποφασίσει. Η δική μα μέχρι τώρα νομική εκτίμηση ποια είναι. ακούστηκε TFTP, PNA, τα άλλα εργαλεία που έχουμε για τη συλλογή στοιχείων είναι πιο περιορισμένα ως προς το πεδίο εφαρμογής και δεν είναι αυτόματο ε, να καταργηθούν αυτά και να ακυρωθούν επειδή ακυρώθηκε η οδηγία ως μια αναλογική. Για κάποια συστήματα PNA στην Ευρώπη ή συστήματα εισόδου-εξόδου που δεν έχουν ακόμα θεσμιστεί, μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από τις συστάσεις της απόφασης του δικαστηρίου, αλλά οι νομικοί μας επαναλαμβάνω εμπειρογνώμονες δεν βλέπουν εδώ καμία σύνδεση της οδηγίας αυτής με άλλα μέσα και εργαλεία που ισχύουν, που είναι πολύ περιορισμένα. Αυτά. Κυρία Πρόεδρε. Έχουμε μόνο 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Έχει κλείσει ο κατάλογος ε, ομιλητών. Εάν υπάρχουν άλλα θέματα μπορείτε να τα υποβάλλετε γραπτός προς την κυρία Μάλμστρομ. Ο κύριος Ράντεφ έχει το λόγο για ένα λεπτό, γιατί έχουμε 20 ομιλητές. Κυρία Επίτροπε, κυρία Μάλστρομ, ε, θα ήθελα ε, να σας πω ότι εδώ και καιρό έχουμε στη Συρία ένα πραγματικά εμφύλιο πόλεμο. Британец, който уби американския журналист Фоли, е само един пример. Тези чуждестранни бойци, както се наричани, неименуемо се връщат. Ме пола ε, παραδείγματα ξένων μαχητών που επιστρέφουν στην Ευρώπη. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω Europol έτσι ώστε να μην ζήσουμε μια άλλη τρομοκρατική δράση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δύο εκατομμύρια πρόσφυγες φεύγουν από το Ιράκ για να σώσουν ε, τη ζωή τους. Έχουμε λοιπόν αυτό το κύμα μεταναστών. Ποια μέτρα θα λάβουμε για να βοηθήσουμε τα, τους ανθρώπους αυτούς να είμαστε δηλαδή ένας φράκτης. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ σε σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την οδηγία ε, σε σχέση με την παρακράτηση και την διατήρηση προσωπικών στοιχείων, νομίζω ότι ε, μιλάμε για τηλεφωνικά στοιχεία και νομίζω ότι είναι πολύ περιοριστική η απόφαση. Το δικαστήριο μιλά για παρακράτηση στοιχείων που δεν είναι συμβατή με το άρθρο 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αν δεν υπάρχει κάποια σαφής υποψία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να έχουμε διατήρηση στοιχείων με την υποψία ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι αναλογικό ή αναγκαίο. Το θέμα όμως παραμένει ανοιχτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όμως ε, δεν ξέρουμε πάντα αν η υποψία είναι βάσιμη, δηλαδή αυτό δεν συμβαδίζει με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν μπορείτε να μην λάβετε υπόψη αυτό τον κίνδυνο, διότι μέσα στα πλαίσια του PNR ή του SWIFT θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η παρακράτηση δεδομένων, η διατήρηση δεδομένων είναι κάτι το οποίο δεν υπερβαίνει ορισμένα χρονικά όρια. Πώς θεωρείτε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του δικαστηρίου. Eh, Ευχαριστώ. Ε, έχετε ήδη απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα που είχα, αλλά τέλος πάντων θα θέσω κάποια άλλα. Σεσίλια, ε, για τις ε, νόμιμες οδούς για να φτάσει κανείς στην Ευρώπη συχνά. Και θέλω να σε ρωτήσω, ε, θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε πρεσβείες, ε, προξενία στις ε, χώρες και ποιος θα μπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις, ποιος θα αποφασίζει πώς πόσοι μπορούν ε, να έρθουν στην Ευρώπη. Ε, και όταν φτάσει κάποιος ε, στη Σουηδία, οι περισσότεροι στη συνέχεια έχουν και άδεια διαμονής. Και έχουμε ήδη αρκετούς που έρχονται στη Σουηδία. Πώς θα γίνει αυτό αν έρχονται ακόμη, περισσότερο, ακόμη περισσότεροι. Και στη συνέχεια είπες ότι και κάποια άλλα κράτη πρέπει να κάνουν προσπάθειες. Τι θα γίνει με ποσοστώσεις, θα το κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποφασίζει πόσοι θα μπαίνουν σε κάθε χώρα εγώ δεν συμφωνώ. Ευχαριστώ ε, η κυρία Ιντβελτ. Ε, νομίζω, νομίζω ότι είπατε το όνομά μου, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ωραία, εγώ είμαι. Λοιπόν, ευχαριστώ ε, που ήρθατε για να συζητήσουμε. Επίτροπε, ε, για την ε, διατήρηση των δεδομένων έχω κάποιε ερωτήσει. Όπω και ο Γιάννα Αλμπρέχτ, ε, πιστεύω ότι πέρα από την διατήρηση υπάρχουν σοβαρότερες επιπτώσεις. Επηρεάζουν το PNR, το TFTP και άλλα παρεμφερή προγράμματα. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει να προωθεί το PNR, ενώ εμείς με ξεκάθαρη πλειοψηφία το απορρίψαμε. Είπαμε δεν θέλουμε. Ε, υπάρχουν και άλλες προτάσεις ε, για την ε, μητρική άδεια παραδείγματος χάρη. Μας είπατε α δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε γιατί δεν έχουμε υποστήριξη στο Συμβούλιο. Ε, λοιπόν τώρα που δεν έχετε υποστήριξη από το Συμβούλιο και από, από νομικής πλευράς δεν ευσταθεί αυτή η πρόταση γιατί επιμένετε με το PNR. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όλα τα σκάνδαλα με τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές και σε σχέση με τις ΕΠΑ και άλλες, ε, με μαζική παρακολούθηση και υποκλοπή, ε, το IC Reach, ε, μια βάση δεδομένων που οι υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου των ήπα μπορούν να ανατρέχουν σε όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί και σαν να είναι Google ψάχνουν και βρίσκουν ό,τι θέλουν. Τι έχετε να πείτε. Και κάτι άλλο, το, τα opt-backins του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάζει τις προτάσεις τον ε, τον οποίο ε, θα διαβουλευτεί το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους. Γιατί δεν μας λέτε μας τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα διαθεσμικά ζητήματα. Η Σιλβίκη Γιώμ ναι, ε, νωρίτερα αναφερθήκατε σε πάρα πολλά και διαφορετικά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα. Εγώ για το θέμα της μετανάστευσης ε, είμαι πεπισμένη ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα στις διάφορες δράσεις, ούτως ώστε να πετυχαίνουν αυτές οι ολιστικές, όπως τις λέμε, προσεγγίσεις. Εγώ τάσουμε πάντα υπέρ μιας σφαιρικής προσέγγισης. Μετά από πέντε χρόνια, και αφού έχετε περάσει από το Κοινοβούλιο, εσείς τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι είναι σφαιρική, οριζόντια, εγκάρσια και συνεκτική προσέγγιση ή αυταπατώμεθα. Ευχαριστούμε, Dali. Ευχαριστώ εντάχει θα ήθελα να μπορούσα να σας μιλήσω στα Μαλτέζικα, ε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν και είδα ότι αυτό ισχύει και σε άλλες επιτροπές. Δεν καλύπτεται η γλώσσα μου. Θα ήθελα να σας πω κύριε Επίτροπε, να σας ε, πω και να σας προτρέψω να ληφθούν μέτρα στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Έχουν ε, γίνει ορισμένα βήματα, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, ιδιαίτερα όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα επιμερισμού ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθίσταται σαφές ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τη Frontex Plus ο Νοέμβριος είναι πρώτον πυλών και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, για την αποστολή της Frontex Plus. Ε, ποιοι κανόνες θα τη διέπουν, ποια θα είναι η γεωγραφική της ε, κάλυψη και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το Mare Nostrum, το οποίο θα έχει πολύ πιο περιορισμένη εμβέλεια Είπατε ότι πολύ λιγότερα κράτη αναλαμβάνουν τους ετούντες άσυλο. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί πρόκειται για θέμα ευρωπαϊκής εμβέλειας. Η κυρία Άτκινσον. Δύο ερωτήματα ως προς την παράνομη μετανόστευση. Το λιμάνι του Ντόβερ είναι στη δική μου εκλογική περιφέρεια και σήμερα ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Καλέ είπε ότι θα κάνει έναν αποκλεισμό του λιμανιού. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση με το ένταλμα κράτησης. Ξέρετε ότι έγινε μία μια παράνομη ε, κράτηση μιας οικογένειας η οποία αφορούσε μια οικογένεια που απλώς ε, πήγε το παιδί της ε, σε μια άλλη χώρα για ιατρική παρακολούθηση. Στη χώρα μου υπήρχε το habeas corpus και θα ήθελα να ρωτήσω πώς λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες, ιδιαίτερα για μια χώρα που έχει αυτό το ιστορικό, αυτή την ιστορία πίσω της. Συμμερίζομαι τα θετικά σχόλια για την εργασία σας και χαίρομαι που θα διοριστείτε εκ νέου. Ως προς το έμπολα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο βιολογικό τομέα. Η Επιτροπή δεν έχει αντιδράσει επαρκώς. Χρειάζεται συνέργεια που δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ως προς τη διαφθορά είπατε ότι η καταπολέμησή της είναι ζωτικής ε, σημασίας. Θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχουν άνθρωποι που ε, καταδικάζουν τη, την Γερμανία ε, σε σχέση με ένα δικαστήριο του Μονάχου που έλαβε αποφάσεις για, τα, για ελληνικά ε, υποβρύχια και πορτογαλικά. Και το δικαιοδοτικό σύστημα της Πορτογαλίας ζητούσε όλα τα, όλες τις λεπτομέρειες της γερμανικής απόφασης, αλλά δεν τα έλαβε. Δηλαδή, αν υπήρξε διαφορά, πού έγινε. Πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει και θα ήθελα τα σχόλιά σας. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Η κυρία Σαρχεντίνη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σύντομα ερωτήσεις. Πρώτον, ε, βασιζόμενοι στο σχόλιο σας, ότι ο κόσμος μπαίνει σε αυτά στις βάρκες ε, γιατί δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σημειώνω. Ελπίζω να ξαναγίνετε επίτροπος με το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Ε, μπορείτε να προβλέψετε κάτι άλλο για την ε, μετανάστευση εργαζομένων ε, την νόμιμη μετανάστευση, γιατί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νομοθεσία για ανειδίκευτούς, για, για χαμηλόβιστους. Ε, επίσης, σύντομα, μάλλον πρόσφατα υπεγράφει η συμφωνία ε, με τον Καναδά για το PNR και είδαμε και την απόφαση του δικαστηρίου για την ε, αποθήκευση και ε, διατήρηση δεδομένων. Μήπως θα πρέπει να προσφύγουμε και εμείς στο δικαστήριο γιατί παραβιάζεται η ίδια μας η νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Σαρσεντίνη, κυρία Χουισμένοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα και πάλι να σας επιστήσω την προσοχή ε, για τις μεταναστευτικές ροές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Στατιστική Υπηρεσία, ε, για το 2014, 7.140 ε, ζήτησαν προστασία ε, στο μεταξύ επίσης άλλες 4.000 και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός αυτός. Καταβάλει προσπάθειες η Βουλγαρία να ε, γιάται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των προσώπων αυτών, αλλά αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες ε, και οικονομικές για να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρόλο μας. Η Βουλγαρία δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Πολλά κράτη-μέλη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε σε κάποιες δυσκολίες από το κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, έχοντας υπόψη πάντα την αρχή της αλληλεγγύης αλλά και της ευθύνης, καθώς επίσης και την οικονομική συμμετοχή ορισμένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε εξακολουθώ να θεωρώ παράλογο που η Επίτροπος βλέπει τη μεταναστευτική πίεση ως ευκαιρία για τη Frontex. Ε, είναι πολύ σαφής η κατάσταση. Έχω δύο ερωτήσεις. Το Frontex Plus τώρα ε, θα είναι συνοριοφύλακες και σε ποια περιοχή θα γίνει αυτό. Ε, και επίσης Πώς θα, γίνεται κάποια καταγραφή, θα σημειώνονται τα στοιχεία όταν θα φτάνουν οι μετανάστες στην Ένωση. Η Βάιτεν, ο κύριος, συγγνώμη, Βάιτεν Χάουζερ, αν το λέω σωστό κιόλας. Ναι, Βάιντεν Χόλτσαρ και κύριος. Äh, κυρία Επιτροπέ, σωστά αναφερθήκατε στο πρόβλημα των ξένων μαχητών foreign fighters γιατί νομίζω ότι είναι πολύ κοντόφθαλμο αν μιλάμε μόνο για απαγόρευση εξόδου ή εισόδου. Δεν ε, λύνονται τα προβλήματα έτσι, ούτε πανάκια είναι. Και δεν θα πρέπει να αποδυναμώνουμε το πρόβλημα ή να το αεροποιούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στρατολόγησης και αφορά πολλούς ε, από κάποιες κοινωνικές ομάδες ε, που γίνονται τσιχαντιστές. Ε, και τομείς ε, που δεν πιστεύει κανείς ότι προέρχονται από τέτοιες τάξεις. Ε, και μάλιστα σε δημόσιους χώρους με πολύ σύγχρονους τρόπους στρατολογούνται, με πάρα πολύ ύπουλους τρόπους και μήπως θα μπορούσαμε να επιμείνουμε πάρα πολύ περισσότερο στην πρόληψη να σπάσουμε αυτά τα πρότυπα και τα σχήματα στρατολόγησης και όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριε Βάιντεν Χόλτσερ. Η κυρία Γκέντς. Δεν κατάλαβα ότι αναφερόσασταν σε μένα. Πολλά ήδη προελέχθησαν, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρεμ γιατί έχουμε μία κοινή πορεία σε αυτά τα θέματα. Εσείς ήσασταν ιδιαίτερα σαφείς. Είπε, είπατε ότι το Mare Nostrum και το Frontex είναι δύο διαφορετικά κα ε, εγχειρήματα και δεν θα υπάρξει αντικατάσταση του ενός από το άλλο. Όπως είπε η Σιλβή είναι δυνατόν να μην προωθήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, γιατί να μην διευρύνουμε το Συμβούλιο Γκάι και να... Το Συμβούλιο Τζάι ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης έτσι ώστε να προβάλλει μία πιο ολιστική πολιτική, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μία εκστρατεία ε, επί του θέματος. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τον έλεγχο των σύνορων, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, όπως έχουν, ε, όπως έχουν πει και πολλοί νομπελίστες ειρήνης ανά τα χρόνια. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες της κυρίας Κένς Γι' αυτό θα ήθελα να ε, πω ορισμένα μόνο πράγματα. Έπλεξε το εγκόμιο στο Μάρε Nostrum, το οποίο έσωσε πολλές ανθρώπινες ε, ζωές, αλλά βλέπουμε ότι αντιστρέφονται τα πράγματα. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ε, πρωτοβουλίες, το Mare Nostrum και το Frontex Plus, με διαφορετικές αρμοδιότητες. Στην ουσία το Frontex Plus θα ασχοληθεί με την εποπτεία και τον έλεγχο των συνόρων και όχι τη διάσωση των ανθρώπινων ζώων. Το πρόβλημα, Επίτροπε, είναι ότι η Ιταλική κυβέρνηση που έδωσε πνοή στο Mare Nostrum δεν λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Το Frontex Plus θα αποτελέσει μια υπέρβαση του Mare Αυτό μας λέει. Άρα κατά τη γνώμη μου και μάλλον και κατά τη δική σας θα αποτελέσει στην ουσία ε, κατάργηση του Mare με πολλούς πνιγμούς της θάλασσες. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, φέτος, το 2014 μόνο, 1.880 άνθρωποι πνίγηκαν στην Ευρώπη προσπαθώντας να διαφύγουν από τη φτώχεια, την πείνα και τους πολέμους που ε, προκαλούν στις χώρες του Νότου οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα συμφέροντα του Βορρά. Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη κάθε χρόνο που την έχετε κάνει φρούριο. Ούτε από το Frontex, ούτε από το Frontex Plus περνάει η λύση. Αλλά από το να σταματήσουμε, πούμε, να πουλάμε όπλα σε χώρες σε εμπόλεμη σύραξη ή να σταματήσουν οι επιχειρήσεις μας να ε, εξακολουθούν να ε, κάνουν ένα πλιάτσικο στις χώρες του Νότου. Ποια είναι η κατάσταση ε, των ε, νοτίων συνόρων στην Σέουτα και Μελίγια που ε, συστηματικά παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ξέρετε ότι δεν τηρείται ευρωπαϊκή και ισπανική νομοθεσία με παράνομες απελάσεις και αποθήσεις. Ποιες είναι οι δυνατότητες να προσφεύγει κανείς σε διεθνή προστασία. Η οργάνωση Human Rights Watch έχει καταγγείλει ε, παραβιάσεις και καταχρήσεις της Ισπανικής χωροφυλακής στη Μελίγια. Αυτή την Ευρώπη θέλετε εσείς. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, λέει η κυρία Λοριστίνα. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά της κυρίας Ε, Ορισμένες φορές φαίνεται ότι δεν υπάρχει και ελπίδα. Δύσκολα τα καθήκοντά της και συγχαρητήρια. Πάντως πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ποια είναι τα δυσκολότερα ζητήματα και πιο σημαντικό ακόμη, έχετε νέες ιδέες για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα για τα οποία δεν είχατε χρόνο ή πόρους. Για την επόμενη επιτροπή ε, ποιοι μπορεί να είναι οι μηχανισμοί, όχι μόνο διάσωση, τι κάνουμε με του ανθρώπου που έρχονται, πώ εντάσσονται, πώ θα ενσωματωθούν ε, στη κοινωνία των κρατών μελών διοχετεύονται κονδύλια ε, σε αυτούς τους μηχανισμούς αλλά συχνά ε, υπάρχουν φόβοι ότι δεν είναι αποτελεσματικοί. Η εκπαίδευσή τους, η παιδεία μετά αυτή γίνεται κυρίως για τα παιδιά και τους νέους. Χρειαζόμαστε μήπως αποτελεσματικότερες πανευρωπαϊκές λύσεις για τα παιδιά πρόσφυγες, για τα παιδιά των προσφύγων. Αντίθετα με αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής, ε, η δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών που γίνονται ένα βάρος, λένε κάποιοι, για την Ευρώπη, όχι, αυτό ε, σημαίνει ότι εμείς αποτύχαμε να τους ενσωματώσουμε. Υπάρχουν ελπίδες για την επόμενη επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ε, ε, κυρία Αντατή. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ακούσαμε κέρια ερωτήματα, ε, δεν θα επανέλθω σε αυτά, όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι κάτι που σχετίζεται με την οργάνωση και αναφερθήκατε σε αυτό και εσείς. Μιλήσατε για τις δυσκολίες χειρισμού των δραστηρικών ροών και των επιπτώσεών τους που τελικά συνιστούν ε, αυτές καθ' αυτές σε προκλήσεις. Δεν σχετίζονται πλέον με τις μεταναστευτικές ροές ως προς την ασφάλεια, ως προς την υγιεινή έμπολα, κάποιο αναφέρθηκε σε αυτό το πρόβλημα. Εμπορία ε, ανθρώπων ε, ε, οργανωμένη εγκληματικότητα. Ε, ε, χρειάζεται ολοένα και στενότερος έλεγχος λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Και πάλι εχθές, παραδείγματος χάρη, στο Καλέ, ο Δήμαρχος μίλησε για αυτό το πρόβλημα, διότι είναι σοβαρές οι επιπτώσεις. Η αύξηση είναι πάνω 50% σε λίγους μόνο μήνες των παρνόμενων μεταναστών, διότι περνάνε από το Καλέ για να πάνε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει ε, ενώπιον αυτών των καταστροφών, διότι οι λαθρομετανάστες ε, τελικά έρχονται διότι, παραδείγματος χάρη στη Μεσογειακή, λέγανε δεν είναι σωστή η διαχείριση και μετά μετατοπίζονται και πάνε στο καλέ μετά την καταστροφή ε, της ε, Λαμπεντούσα, γιατί μόνο τους, στόχου είναι να πάνε σε ένα κράτος μέλο και στην προκειμένη περίπτωση θέλουν να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, το Frontex Ναι, θα έχει μια επίπτωση για τον περιορισμό της λαθρέα μετανάστευση και ελπίζω και την ε, αποκλιμάκωση αυτών των ε, ανθρώπινων τραγωδιών που βιώνουμε, ε, πώς θα ενισχύσουμε την ε, ε, πάταξη της λαθρές μετανάστευσης που παρά τις ε, προσπάθειές μας τελικά εκφεύγουν των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων και εισέρχονται στο χώρο Σέγγεν. Για την υποστήριξη για το Frontex ΣΥΝ αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης γιατί το ξεχνάμε συχνά αυτό ε, σήμανση, καλύτερη σήμανση δακτυλικά αποτυπώματα. κυρία Ντάτη, ξέρετε, έχουμε άλλους τρεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα ολοκληρώσω. Θέλω να ξέρω αν θα υπάρξει χαρτοφυλάκιο. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην προεκλογική του μας είπε, και υπενθυμίζω ότι και νικήσαμε, ότι θα υπάρχει ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο. Ισχύει. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω το λόγο ή όχι, ο κύριος Μπέκερ. Α, όχι, ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, για την εκτενέστατη απάντηση και εξήγηση για πολλά θέματα και δύσκολα προβλήματα. Μια ερώτηση έχω μόνο. Πώς μπορεί κανείς να καταφέρει... Ε, ε, να ολοκληρωθεί το PNR από το Συμβούλιο και να αρχίσει ήδη εντός του 2015 ο τριμερής διάλογος. Δεν είναι ξεκάθαρο. Κάποια κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα και δεν είναι και πρόθυμα να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Εσείς πώς το αξιολογείτε και πώς το βλέπετε και τι προτίθεστε να κάνετε για να ε, δρομολογηθεί καλύτερα αυτή η διαδικασία. Αν θέλετε να το πω κιόλας, να πιέσετε την Προεδρία για να παρουσιάσουν μία ατζέντα στην κοινή γνώμη για το πώς προτίθεται να διαχειριστούν όλη αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα τρεις, παρακαλώ. Post, Bild και Μπέκερ. Και τελευταία κυρία Ζίπελ, για ένα λεπτάκι μόνο. Σας παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Μέχρι τις 4 προβλεπόταν, άντε πέντε λεπτά ακόμα. Για να ακούσουμε και την κυρία Επίτροπο. Eh, Ευχαριστώ. Ε, έχοντας ακούσει τώρα τις ε, συζητήσει που έγιναν ε, για αυτά τα θέματα, νιώθω ότι είναι πάρα νιώθω μια δυσφορία, μια δυσαρέσκεια σε σχέση με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι είναι ο χειρό τελικά η Ευρώπη, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Frontex είναι μας είπατε, εγώ ήλπιζα ότι θα αντικαθιστούσε το Mare Νόμιζα ότι αυτή ήταν η πρόθεση ε, και όταν μιλάμε για τους ε, οικονομικούς πόρους, ε, για την διάσωση, γιατί αυτό έκανε η επιχείρηση Μαρενόστρουμ, μας λένε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν πόρους για να αναλάβουν τα έξω μια τέτοια οργάνωση και τα αφήσαμε μόνο στην Ιταλία. Μόνο η Ιταλία είχε λεφτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια για να αντιμετωπίσει μια κοινή απειλή ε, στο κάτω-κάτω της γραφής. Ε, είναι σκάνδαλο αυτό. Τελικά, ε, εμείς αυτά που, αυτές τις αρχές που έχουμε στο χαρτί τις υπερασπιζόμαστε στην πράξη. Ευχαριστώ, κυρία Μπίλτ, ευχαριστώ. Ε, Επίτροπε, ε, συγχαρητήρια για το διορισμό σας. Ε, όπως και οι συνάδελφοι, θέλω και εγώ να ασχοληθούμε με τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, βλέποντας το τι γίνεται στη Μεσόγειο. Χαίρομαι που εξακολουθείτε να έχετε τη δέσμευση κοινή ευθύνη ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Σουηδία υποδέχεται 21% των ε, προσφύγων ε, που εισέρχονται στην Ευρώπη. Δεν μιλάμε μόνο για την κατάσταση στην Μεσόγειο. Ο στόχο είναι να σώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και περνάνε ολόκληρη τη ζωή του στην Σουηδία και αυτή η πρόκληση είναι διαφορετική φύση και χαίρομαι που ασχολείστε και με την περίοδο μετά την υποδοχή των για την εμπορία. Τι σκοπεύετε να κάνετε ούτως ώστε ε, τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, τις οδηγίες και τους κανονισμούς που εγκρίναμε στην προηγούμενη θητεία για τη στρατηγική τώρα που έχουμε για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ε, μία από τις αποφάσεις που λάβαμε, ε, τι θα γίνει, θα εκπνεύσει το σχέδιο δράσης, ε, θα συντάξετε νέο σχέδιο δράσης για να αναδειχθούν τα παιδιά σε προτεραιότητα. Ευχαριστούμε κυρία Μπέλη, τον κύριο Μπέκερ. Ευχαριστώ. Ζήτησα πολύ νωρίς το λόγο, πάλι καλά που μου τον δώσατε. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε κύρια Επίτροπε. Οκταπλασιάστηκε η μετανάστευση σε αριθμούς από τη Μεσόγειο και είναι σαφές ότι είναι τελείως ανεπαρκής ο προϋπολογισμός του Frontex. Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω να αυξηθούν τα ποσά κατά 20 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω να ε, συμφωνήσουν και οι αρμόδιοι. Εσείς πώς βλέπετε το προπολογισμό της Frontex για το 2015. Δεύτερο, μιλήσατε για τους ξένους μαχητές και είπατε ότι εκπονείται με ΑΙ αυτή τη στιγμή ε, μια νέα πρόταση. Για πότε. Τρίτη ερώτηση για τη μετανάστευση γενικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται να ε, ασχοληθεί και με άλλους τομείς πολιτικής, ας πούμε η συνεργασία με τις τρίτες χώρες να βελτιωθεί εκεί. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Τελευταία η κυρία Ζίπελ, δεύτερη φορά αλλά για πολύ λίγο παρακαλώ. Ναι, ναι, πολύ λίγο. Για το θέμα αυτό του Frontex, η Ιταλία ε, δήλωσε ότι τερματίζει ε, το πρόγραμμα Mare Nostrum και θα αναλάβει Frontex, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν δύναται. Λοιπόν, τι έχετε συμφωνήσει συγκεκριμένα με τον κύριο Αλφάνο. Δεν θέλω να σας δυσκολεύσω την απάντηση, αλλά ο Ιταλός Υπουργός είδαμε τώρα μόλις να δηλώνει και παρακαλώ να μας το επιβεβαιώσετε ότι θα συνεχίσει το Μάρε Νόστρομ στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας και από εκεί και πέρα στα διεθνή ύδατα θα αναλάβει η Frontex. Τι έχετε να απαντήσετε εδώ. Παρακαλώ κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο σύντομα γιατί έχουμε και ψηφοφορίες και μάλιστα τον προπολογισμό. Βεβαίως θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά είχαμε πολλές ε, ερωτήσεις. Κυρία Ντατή, το κατά πόσο θα υπάρξει επίτροπος που θα ασχοληθεί μόνο με το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, δεν το ξέρω. Ο πρόεδρος Γιούνκερ θα ασχοληθεί με τα χαρτοφυλάκια και νομίζω την επόμενη εβδομάδα όλα θα είναι έτοιμα Μπορείτε να του υποβάλλετε το ερώτημα την επόμενη εβδομάδα. Υποβλήθηκαν πολλές ε, ερωτήσεις που καλύπτουν το θέμα ε, της δικαιοσύνης. Γι' αυτό θα αφήσω σε άλλους συναδέλφους το θέμα του εντάλματος, όπου το Συμβούλιο ε, ακολουθεί βραδύτα τους ρυθμούς. Τώρα ως προς τη μετανάστευση γιατί πολλοί ρωτήσατε, με αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος. Όχι, πέρα από θέματα, ε, τα θέματα της οικονομίας, η μετανάστευση είναι το δεύτερο μείζον ζήτημα στην Ευρώπη. Η μετανάστευση είναι ένα διεθνές ε, φαινόμενο. Όλοι, πολλοί μάλλον, αποζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Άλλοι θέλουν να διαφύγουν από την καταστολή, από πολέμους, από την φτώχεια και από το λοιμό, όπως βλέπουμε στη Συρία και αλλού. Ε, ένα μικρό μέρος αυτών θα προσέλθουν στην Ευρώπη. 100.000 μόνο στην Ευρώπη από τα τρία εκατομμύρια και τα 6 εκατομμύρια συνολικά. Βεβαίως και από το Ιράκ θα προσέλθουν. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όποτε μπορούμε, αλλά να γνωρίζουμε ότι έχουμε δεσμεύσεις και αξίες. Βεβαίως όλοι αυτοί δεν θα έρθουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να διαχειριστούμε την παράνομη μετανάστευση, την μετανάστευση χορήγησης ασύλου και την ε, οικονομική μετανάστευση. Προσπαθούμε να έχουμε μία συνολική εικόνα, διότι σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική, με το εμπόριο και ούτω καθεξής. Ελπίζω η νέα Επιτροπή να συνεισφέρει καθώς και το ε, Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μη σκεφτόσαστε με στεγανά. Υπάρχουν πολλές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που το αντιμετωπίζουν ως απειλή. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, αλλά είναι μια πραγματικότητα θα πρέπει να δούμε πώς χειρίζονται το θέμα αυτό κυβερνήσεις, κόμματα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να έχουμε συνεκτική προσέγγιση από το σημείο όπου εκτοπίζονται αυτοί οι άνθρωποι μέχρι ότου έρθουν σε μας. Η Frontex Plus δεν είναι μία αντικατάσταση του ε, Κυρία Σίμπελ, δεν μπορώ να το ε, σχολιώσω, γιατί δεν ξέρω τι είπε ο Υπουργός σήμερα. Είναι Ιταλικό θέμα. Εμείς θα συμπληρώσουμε αυτή την εργασία, αλλά δεν αντικαθίσταται θα είναι πιο περιερισμένη η εμβέλεια αυτού του εγχειρήματος που προβάλλουμε τώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και περισσότερες δεσμεύσεις και από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε και οι 28 χώρες να πούν ότι ναι, ο καθένας θα κάνει το δικό του. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να το κάνουν, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε από τα 28 κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν υπάρχει νόμος ε, για να επιβάλλουμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε έκκληση μόνο με βάση τις ευρωπαϊκές συμβάσεις ως προς την οικονομική μετανάστευση και την μετανάστευση εργασίας. Θα ήθελα να είχαμε περισσότερους κανόνες. Κυρία Βίκστρομ, ξέρετε πάρα πολύ δύσκολο πώς είναι δυνατόν να περάσει η οδηγία για την έρευνα. Ήδη αυτή δεν μπορεί να εγκριθεί εύκολα. Το Συμβούλιο δυσχεραίνει τη θέση μας, άρα θα είναι δύσκολο να προβάλλουμε νέα νομοθεσία, αλλά προωθούμε περισσότερο διάλογο, να δούμε τις δεξιότητες, το δημογραφικό και ελπίζω όποιος αναλάβει το χαρτοφυλάκιο να το αντιμετωπίσει. Για το έμπολα θα ήθελα να πω ότι δύο ε, επίτροποι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Κάναμε πολλά και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με δίκτυα, με γιατρούς, δίνουμε χρήματα για την επιδημία αυτή. Είναι μια πολύ σοβαρή νόσος και δεν υπάρχει κίνδυνος για την Ευρώπη, αλλά το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς. Αν ρωτήσετε τους συναδέλφους στην Επιτροπή Υγείας, μάλλον Γενική Διεύθυνση για την Υγεία και η ΑΦΕΤ, On the Ebola uh, issue. Η Επιτροπή Υγείας θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, PNR και οδηγία για την διατήρηση στοιχείων. Είναι δύσκολο. Πολύ γνωρίζετε ότι η οδηγία παρακράτησης στοιχείων δεν με βρήκε σύμφωνη, αλλά θα πρέπει να πω ότι είχαμε να κάνουμε με μία συσσόρευση στοιχείων. Το PNR αφορά πληροφορίες που εγώ δίνω ως επιβάτης στον αερομεταφορέα. Είναι κάτι το διαφορετικό. Όμως ε, οι νομικοί εμπειρογνώμονες ασχολούνται με το θέμα έτσι ώστε να γίνει μια αξιολόγηση, ειδικά τις συμφωνίες PNR. Τώρα, γιατί ασχολούμαστε περισσότερο και ιδιαίτερα με το PNR. Έχω την ε, εντύπωση ότι αναπέμψατε το ζήτημα στην Επιτροπή. Δεν το έχετε απορρίψει το νέο PNR και 14 χώρες έχουν ένα εθνικό σύστημα PNR. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, PNR έτσι ώστε να έχουμε μια συγκεκριμένη εμβέλεια προστασίας και ρύθμισης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό να μας απασχολήσει περαιτέρω. Για τους ξένους μαχητές σας είπα ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τα κράτη-μέλη. Εμείς δεν προτείνουμε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά προβαίνουμε σε ανταλλαγή απόψεων και προβάλλουμε και προγράμματα πρόληψης. Υπάρχουν ε, προγράμματα εξόδου όχι μόνο για τους ξένους μαχητές, αλλά και για τους εξτρεμιστές οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν από αυτό το βίο περιβάλλον και έχουμε στοιχεία γιατί πρόκειται για δραστηριότητες που μας απασχολούν. Μας απασχολεί και το χρηματοδοτικό πλαίσιο, αλλά το πλαίσιο καταστολής αφορά το εθνικό καθαρά επίπεδο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην ε, ξέχασα κάτι. Α, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Αν ναι, ξέχασα. Ξέχασα μια στιγμή. Το άρθρο 36, πολύ σημαντικό, αυτό θέλατε να ρωτήσετε. Για το opt-in και opt-out της Βρετανίας. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις κάνει και το Συμβούλιο δέχεται να έρθει κάποιος αρμόδιος να σας ενημερώσει από την αρμόδια γενική διεύθυνση. Συνεννοηθείτε παρακαλώ με τη γραμματεία για να ενημερωθείτε. Η κυρία Ενιτφέλτ. Ναι, ευχαριστώ για την απάντηση αυτή. Ε, έχω καταλάβει ότι έχετε στείλει στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου μια ενημερωτική επιστολή. Καλό θα ήταν να τη λάβουν και οι ευρωβουλευτές την ίδια ενημέρωση, όχι μόνο γενικώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλή τύχη στις εκλογές και θα τα ξαναπούμε άλλη μια φορά πριν λήξει η θητεία σας φαντάζομαι. Στο καλό να πάτε. Ε, euh, λοιπόν, συνεχίζουμε και ψηφίζουμε κιόλα. Κύριε Σιγητά, θέλετε το λόγο? Παρακαλώ. Όχι? Αν δεν θέλετε να λάβετε το λόγο λοιπόν, θα σας δώσω δύο λεπτά ε, διάλειμμα λίγο να ανασυνταχθούμε για να ψηφίσουμε. Μάκου καφέ από τον Είμαστε Je vous en prie, on va continuer avec le vote. Ε, θα πρέπει να αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ, καθίστε και ησυχία. Chers collègues, on va continuer avec le vote, mais après... Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Madame Bild, je vous en prie. Je vous en prie de tester d'abord les cartes électroniques. Παρακαλώ βγάλτε τις ηλεκτρονικές κάρτες σας για την ψηφοφορία. Est-ce que tout le monde a posé les cartes déjà? Έχετε τις κάρτες σας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Βλέπουμε ότι λειτουργεί. Και ο αριθμός των ομάδων... Ναι, ναι, τεστ ήταν αυτό. Θα αρχίσουμε τώρα με τις ε, τροπολογίες που έχουν ήδη κατατεθεί.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 24 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι χρειάζεται ηλεκτρονική εξακρίβωση. Λοιπόν, επαλήθευση ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Le vote est clos maintenant. Le... Πέρας. Απορρίπτεται, λέει η πρόεδρος. Παρακαλώ να, να επαναληφθεί η ψηφοφορία. τη λείπανε κάποιες κάρτες. Πέρας. Λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας. Υπάρχουν, ε, υπάρχει και κάποιος άλλος ε, στο μείον, οπότε... Σοψηφία. Απορρίπτεται. Πρόεδρε, ένα λεπτάκι. Γιατί είναι δικιά μου η τροπολογία. Πρώτα ε, πέρασε, δεν ξέρω τι έγινε γιατί δεν το εξηγήσατε, τώρα έχασα, προσθέτετε ψήφους, αφαιρείτε ψήφους, μπορείτε να εξηγήσετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Κυρία Σεντεντίνη, ε, συγγνώμη να σε εξηγήσω. Ε, στους σοσιαλιστές έχουμε άλλον έναν, άλλη μία ψήφο και έχουμε και μία ψήφο μείον. Συγγνώμη, στον πρώτο γύρο ζητήσατε δεύτερο γύρο, χωρίς να μας εξηγήσετε γιατί χρειαζόταν δεύτερος επαναληπτικός. Κανονικά, αν η έκβαση παραμένει η ίδια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν παραπονιέται κανείς, ε, ε όμως τώρα άλλαξε. Ε, πρώτα εγκρίθηκε και μετά απορρίφθηκε και ε, συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνώ με τη διαδικασία. Η γραμματεία ε, μου εξήγησε ότι και στην, στον πρώτο γύρο υπήρχε ισοψηφία γιατί ε, λείπαν οι δύο κάρτες αλλά είχαμε και δύο που ήταν ε, κατά. Και έτσι προέκυψε η ισοψηφία. Δεν έχει γίνει τίποτε άλλο. Θα συνεχίσουμε τώρα με την τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 01. Ε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Διορθώνει η πρόεδρος. 29. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τριάντα. Υπέρ. Η 30, τη 30 ψηφίζουμε. Ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Ε, σχόλια εκτός μικροφώνου, δεν ακούνε οι διερμηνείς δυστυχώς. Ε, συγγνώμη, ε, υπήρξε μια σύγχυση. Ψηφίσαμε για την 30 και για την 32. Εγώ ζητώ επανάληψη της ψηφοφορίας για την 30. Απαντάει η Πρόεδρος για την 32 ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Ε, κατά. Σαρτζεντίνη. Πρόεδρε, ε, η κυρία Ζήπελ ε, κάνει σχόλιο για την 30, δεν απαντήσατε, δεν ψήφισα εγώ για την 32. Συγγνώμη, ε, πρέπει να ξεκαθαρίζεται όταν υπάρχει διαδικαστικό πρόεδρος. Κυρία Σατζεντίνη, έχει απορριφθεί η 30, απερίφθη μετά την ψηφοφορία. Συγγνώμη, ε, αλλά... Μετά ψηφίσαμε για την 32. Ξαναλέω, 32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τριάντα ένα τώρα υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Τριάντα τρία, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μηδέν τριά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 04 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 διορθώνει πρόεδρος 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 06 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 07 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι τροπολογίες 39 και 43 τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Όχι καταπίπτει. Λέει πρόεδρος και η 08 το ίδιο. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. επαλήθευση παρακαλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le vote est clos. Le résultat. Πέρασε. Εγκρίνεται. qui est pour. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 09 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται λέει η πρόεδρο ωραία θα επαληθεύσουμε 54 ψηφίζουμε 54 54. Ψηφίζουμε. Le vote est clos. Le résultat. Πέρας. Και να δούμε και το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε. Τροπολογία 58 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε εντάξει. 63. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Νομίζω ότι είναι σαφές το αποτέλεσμα, αν θέλετε όμως μπορούμε να επαληθεύσουμε. 64 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 και 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 19 τελευταία ε, η οποία καταπίπτει λοιπόν τώρα ψήφισμα τροπολογία 1 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 σε δύο τμήματα επίσης. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 2 υπέρ. Κατά. Νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία συμβασμού 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε, εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα, συνδυασμός 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με συγχωρείτε. Τρεις δεν ψήφισαν. Μπορούμε να ψηφίσουμε άλλη μία φορά σας παρακαλώ, γιατί λείπουν τρεις ψήφοι. Εντάξει. Εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος. La réunion de la Συνέχιση αύριο στις 9.30 λίτη συνεδρίαση.